Δικονομικέ εγγύσει για παιδιά που είναι ύποπτοι κατηγορούμενοι στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών. Δίνω αμέσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε κύριε Γιουρόβα, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή, του Σκιώδης συγητές και τη προεδ... της Προεδρίας, ιδίως Λουξεμβουρού, κατά από τις οποίες έγιναν οι διαπραγματεύσεις για την επικοδομητική εικόνα που είχαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ένα χρόνο έχει που ανέλαβα από την Επιτροπή Λίβε την ευθύνη για την εξέταση του κειμένου της οδηγίας. Ε, η δουλειά στηριζόταν στην επιθυμία να έχουμε μια διάταξη που για πρώτη φορά θα εξέταζε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ανηλίκων σε υπερεθνικό επίκαιο παρέχοντας οικονομικές εγγύησεις για τους ανηλίκους αυτούς. Εννέα τρίλογοι χρειάστηκαν, δύσκολοι σε κάποιες περιπτώσεις και πολλές τεχνικές συναντήσεις πριν φτάσουμε σε μια οριστική συμφωνία που θεωρώ πολύ θετική και όπου μπορώ να υπάρξει συνένεση στο σώμα. Πολύ... Πολλές διαφορές υπάρχουν ακόμα μεταξύ των νομικών συστημάτων και των για την μετώπιση των, των ανηλίκων. Η οδηγία προσπαθεί να καλύψει τις αποκλήσεις αυτές ορίζοντας και εντοπίζοντας ε, σαφή δικαιώματα για τους ε, κατηγορούμενους ή ε, ύποπτους ανηλίκους με υψηλό επίπεδο εγγύσεων. Χρειάστηκε να θέσουμε στο κέντρο το πρωταρχικό συμφέρον του παιδιού που κατοχυρώνεται και στο άρθρο 18 της ε, Ευρωπαϊκής ε, Χάρτας Δικαιωμάτων Ανθρώπου που για πρώτη φορά εισάγεται στην στο ποινικό πλαίσιο. Η προστιθέμενη αξία της ε, οδηγίας έρχεται ακριβώς το ότι δίνει στους ανηλίκους πέραν συγκεκριμένων δικονομικών δικαιωμάτων και μια ειδική αντιμετώπιση λόγω του ειδικού χαρακτήρα του ως ανηλίκων που πρέπει να την, την χάνουν ειδική προστασία. Πολλές είναι οι διατάξεις των, ε, της τι τις οποίες παρεμβαίνει η οδηγία αλλά δεν θα τις χαλιώσω όλες. Θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 6 ωστόσο που προβλέπει το δικαίωμα ανηλίκου να προστατεύεται από έναν ε, έχουν ευθύνη την ε, υπεράσπιση του. Είναι ένα δύσκολο σημείο που με ικανοποιεί συνολικά, διότι περιγράφει περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η συνδρομή συνήγορου για την σωστή εφαρμογή όλων των εγγυήσεων και για να βοηθήσει το παιδί να καταλάβει την πορεία της διαδικασίας στην οποία εμπλέκεται. Για το λόγο αυτό, παρότι μπορούμε να δούμε διάφορες περιπτώσεις παρέκκλησης ανάλογα με την ηλικία του ανηλίκου, το ότι βαρύτητα το αδικήματος και τα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν κατόπιν, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την παρουσία του συνηγόρου από την αρχική φάση των ερευνών, ιδίω όταν ο ανήλικος που εξετάζεται από την αστυνομία είναι σε στέρηση ελευθερίας. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της οδηγίας είναι αυτό που απαιτεί από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τον ανήλικο σε αξιολόγηση που γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό για να υποστηρίξει αποφάσεις για μέτρα προς όφελος του ανηλίκου, για την καταλληλότητα πιθανών, ε, προ, ε, ε, πιθανών μέτρων στέρης ελευθερία και άλλες δραστηριότητε. Επίσης, είναι σημαντική η εκπαίδευση εκείνων που εμπλέκονται στη διαδικασία, ξεκινώντας από τα αστυνομικά όργανα, τους δικαστικούς και τους σύνηγους. Προβλέπεται στην οδηγία ότι αυτοί πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση και πρόσβαση αυτή για να εξασφαλίσουν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επανένταξης του ανηλίκου μετά την ποινική εμπειρία, η κράτηση θεωρείται πάντα ως ε, ε, ακραίο μέσο όταν τα εναλλακτικά μέτρα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικά ή εφαρμοστέα. Όταν πρέπει να στερηθεί η προσωπική, ο ανήλικος της προσωπικής του ελευθερίας πρέπει να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει για να μπορέσει να συνεχίσει την εκπαίδευση και να διατηρηθεί η ψυχοκοινωνική του ισορροπία. Η οδηγία πρέπει για πρώτη φορά να μπορεί να, να σταθεροποιήσει στην Ευρώπη μια παρόμοια αντιμετώπιση των ανηλίκων. Η οδηγία θα πρέπει να πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση για τον ορισμό ενός κοινού μοντέλου δίκαιης δίκης για τους ανηλίκους συμβάλλοντας και στον ε, ποινικό χώρο στη δημιουργία μιας δικαιοσύνης προς όφελος των ανηλίκων. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Γιούροβα. Έχετε το λόγο κυρία Γιώργα. Κυρίες και κύριοι, θα ψηφίσουμε σήμερα για την οδηγία για, τις, για τα μέτρα προστασίας, τα δικονομικά μέτρα προστασίας για τα παιδιά για τα οποία, τα οποία κατηγορούνται στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών είναι σημαντικό γιατί ορίζει συγκεκριμένα δικαιώματα για τα παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικέ διαδικασίες και προστατεύει τα παιδιά αυτά σε όλες τις φάσεις. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε ποινικέ διαδικασίες λόγω της ε, ανοριμότητάς του Ένα εκατομμύριο παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ότι έρχονται σε επαφή με την αστυνομία και τη δικαστική εξουσία σε αιτήσια βάση. Απαιτείται λοιπόν η υψηλότερη δυνατή προστασία. Η οδηγία αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την δημιουργία ενός χώρου δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα επίπεδα προστασίας που προσφέρονται ε, στα παιδιά στις ε, διαδικασίες αυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις το επίπεδο προστασίας είναι ανεπαρκές σε σχέση με τα διεθνή επίπεδα. Η συγκεκριμένη οδηγία λοιπόν αυτή τη στιγμή υιοθετηθεί θα βελτιώσει τις ε, εγγυήσεις αυτές για τα παιδιά όταν αντιμετωπίζουν τις ε, ποινικέ διαδικασίες. Ταυτόχρονα η οδηγία θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη μιας σωστής μορφής δικαιοσύνης για τους νέους. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη για τα παιδιά θα είναι δεδομένο και θα βοηθήσει την κοινωνική τους επανένταξη και θα τα αποτρέψει από το να ξαναδιαπράξουν τις ίδιες ενέργειες. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ την εισηγήτριά σας, την κυρία Κινίτσι, για την προσπάθειά της στην προσωπική της αφοσίωση που κατέστησε δυνατή την συμφωνία μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις. Την ευχαριστώ πολύ. Η κατάληξη των διαπραγματεύσεων είναι ένα σωστά ισορροπημένο κείμενο το οποίο συμφωνεί με την αρχή του άρθρου 24 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ότι τα συμφέροντα των παιδιών θα πρέπει να είναι η κυρίαρχη ανησυχία μας. Ε, τα παιδιά θα ωφεληθούν από την βοήθεια από ε, νομική συμβουλή και προστασία σε όλες τις φάσεις ε, και κάθε φορά που υπάρχει στέρηση της ελευθερίας. Η στέρηση της ελευθερίας δεν μπορεί να επιβληθεί αν το παιδί δεν έχει συνοδευτεί από δικηγόρο εξ αρχής κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν και άλλες μορφές προστασίας όπως η βοήθεια από τους γονείς οι άλλα κατάλληλα πρόσωπα θα έχουν το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικότητάς τους, στην δυνακότητα επίσης διεξαγωγής της δίκης με απουσία του κοινού. Τα παιδιά θα έχουν επίσης το δικαίωμα σε προσωπικές αξιολογήσεις έτσι ώστε οι συγκεκριμένες ανάγκες τους σχετικά με την προστασία, την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη λαμβάνονται πλήρως υπόψη. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανοποιημένη γιατί το έγγραφο προβλέπει ότι οι παιδιά θα πρέπει να κρατούνται ε, ξεχωριστά από τους ε, ενήλικους στα πλαίσια ε, της κράτησής τους πριν από τη δίκη. Η οδηγία αυτή λοιπόν θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίζει τα παιδιά που είναι τα πιο ευάλωτα πρόσωπα που εμπλέκονται σε ποινικέ διαδικασίες και γι' αυτό θα ήθελα να σας δείσω να υπερψηφίσετε την οδηγία αυτή σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζουμε με τον κύριο Τσακή εκ μέρους ε, του ΕΛΚ για 1,5 λεπτό. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Κινίτσι για την έκθεσή τη. και σα ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε. Εκ μέρου του ΕΛΚ χαίρομαι διότι έχουμε μια οδηγία που είναι αποδεκτή και στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη. Κατά τις διαπραγματεύσει. είναι σημαντικό να υπάρχει μια ε, οδηγία εφικτή ε, που να μπορεί να μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο και ελπίζω αύριο να ψηφιστεί αυτό το κείμενο το οποίο δίδει πραγματικά προστασία ε, στους νέους. Θέλουμε να έχουμε ένα νόμο ο οποίος να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε κάποιο κρίσιμο σημείο των διαπραγματεύσεων τονίσαμε τη σημασία που έχει η συνδρομή δικηγόρου. Όταν όμως δεν είναι εφικτό αυτό ε, ε, θα έπρεπε να εξετάσουμε μήπως τυχόν θέτουμε και σε κίνδυνο ε, τα παιδιά όταν απαιτούμε σε κάθε περίπτωση την παρουσία δικηγόρου. Σημαντική είναι η διάταξη ότι θα πρέπει να κρατούνται χωριστά τα παιδιά από τους ενηλίκους θα πρέπει να φροντίσουμε να μην στιγματίζονται τα παιδιά και να φροντίζουμε να γίνεται πιο εύκολη η επανένταξή τους στην κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν πολύ προσεκτικά να χειριστούμε αυτά τα θέματα και η οδηγία αυτή διασφαλίζει αυτά τα οποία επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών, κ. Λόπε Αγγιλάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητούμε εδώ ένα κείμενο σε πρώτη ανάγνωση πολύ σημαντικό που εντάσσεται στο γενικότερο πακέτο δικονομικών εγγύησεων αλλά αφορά μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα τους ανήλικους που είναι το 12% δεν είναι λίγοι το 12% των ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι ή δικάζονται. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή από πλευράς Κοινοβουλίου. Παρέχεται μια εξατομικευμένη προστασία εγί συμμετοχή των ατόμων που έχουν την επιμέλεια του ανηλίκου στις διαδικασίες, ιδίως γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί μόνο στο ως έσχατο μέτρο η κράτηση του ανηλίκου. Επίσης απαιτείται η ιατρική εξέταση του ανηλίκου. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι ότι υλοποιούμε με το κείμενο αυτό το σύνολο των δικονομικών εγγύσεων που είχαν ξεκινήσει με, βάση το, με νομική βάση το άρθρο 32 και με σεβασμό του, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που παρεμβαίνει μόνο από, βάση της αρχής αναλογικότητας βεβαίως και της αρχής αναγκαιότητας. Σας θυμίζω ότι κάθε πράξη δραστηριότητα, κάθε δραστηριότητα ενός ε, της αρχής χωρίς νομιμοποίηση είναι τυραννική δράση. Ο κύριος Τζαμπάσκι. Πρόεδρε Επίτροπε, συνάδελφοι, συγχαίρω την εισηγήτρια και τους χειώδη εισηγητής για, την, ε, για το κείμενο που υλοποιήσαμε, που είναι σημαντικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στον τρόπο προστασίας των δικαιωμάτων των υλίκων από χώρα σε χώρα. Ένα εκατομμύριο παιδιά το χρόνο έρχονται σε επαφή με ε, δικαστήρια ανηλίκων ή την αστυνομία. Είναι ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και χρειάζονται προστασία για το λόγο αυτό. Πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά τις τρύπες που υπάρχουν στα διάφορα ένομα, στις διάφορες ένωμες τάξεις, προσπαθώντας να ο, κάνουμε ομοιόμορφα τα στάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες για αυτούς. Δύο λεπτά, κυρία Γκρισμπέκ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα που η δημοκρατία και το κράτος δικαίου υφίστανται επιθέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ θετικό το να καταφέρουμε να έχουμε μια ωραία συμφωνία για αυτή την οδηγία και μάλιστα διότι αυτή η οδηγία αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, τα παιδιά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ε, κάτι που θέλω να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά σήμερα, ότι τα παιδιά είναι η μελλοντικοί ενήλικοι και αποτελούν το μέλλον μας. Το να δίνουμε λοιπόν προτεραιότητα τα παιδιά μέσα σε αυτό το κείμενο μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε. Ιδιαίτερα Χαιρετίζω την ε, αποφασιστικότητα και την ε, πεισματική δουλειά που έκανε η Κατερίνα Κινίτσι επί μήνες και την ευχαριστώ που κατάφερε να επιτύχει αυτή την ιδιαίτερα φιλόδοξη πρωτοβουλία μαζί με όλους τους συναδέλφους όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα που θεωρούμε θεμελιώδη. Είναι θεμελιώδη διότι η δικαιοσύνη δεν είναι πάντοτε ή πολύ συχνά δεν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών και των νέων. Φανταστείτε την ψυχολογική κατάσταση ενός παιδιού σε ένα περιβάλλον διοκτικών αρχών ή δικαστηρίου. Χρειάζονται λοιπόν τα μέτρα προστασίας, χρειάζεται μια δικαιοσύνη που να είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία των παιδιών και στις ανάγκες τους θα πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά κάτι το οποίο είναι αξιόπιστο και κατανοητό. Χρειάζεται μία προσωπική αξιολόγηση του παιδιού με πρόσβαση σε συνδρομή δικηγόρου και θα πρέπει να αναζητούνται και ως το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ε, ως προς την κράτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους των Πρεσίνων η κυρία Λάμπερτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την οδηγία αυτή, διότι στις διαπραγματεύσεις που έγιναν κράτησε μια ισχυρή και θετική γραμμή. Έχουμε πολύ λίγες παρεκκλήσεις που περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μειώνοντας την ευελιξία την οποία επιζητούσε το Συμβούλιο συχνά. Είναι σημαντικό αυτό το πακέτο για τα δικονομικά δικαιώματα. Νομίζω ότι έχουμε βελτιώσει τα δικαιώματα ε, των παιδιών. Η πρόσβαση σε δικηγόρο είναι βασικό σημείο και η δική μας πολιτική ομάδα ανησυχεί για το άρθρο 6.6 σχετικά με την αναλογικότητα όταν θα εφαρμοστούν αυτά σε εθνικό δίκαιο δεν ξέρουμε πώς θα μεταφερθούν στην πράξη. Πάντω συνολικά η οδηγία αυτή θεωρούμε ότι είναι ένα καλό νομοθετικό εργαλείο που θα βελτιώσει τα δικαιώματα των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέτεν, ένα λεπτό, εκ μέρους του EFT. Ευχαριστώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εγκρίνει αυτή την νομοθεσία για δύο λόγους. Καταρχήν διότι έχουμε opt-out και δεύτερον διότι ήδη έχουμε στο δικό μας δίκαιο τέτοιες εγγύησεις. Φαίνεται ότι κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν βασικές εγγύησεις για τα παιδιά στο νομικό του σύστημα και αυτό πραγματικά μας σοκάρει όπως το δικαίωμα για την εκπροσώπηση από δικηγόρο, όπως το δικαίωμα το παιδί να κρατείται χωριστά από ενηλίκους, το δικαίωμα επίσκεψης από τον γονέα που έχει τη από κάποιο άλλο ενδεδειγμένο ενήλικο. Αυτό πραγματικά μας ε, σοκάρει. Πώς μπορούν άλλα κράτη-μέλη να μην έχουν τέτοια βασικά ε, μέτρα προστασίας. Ε, ε, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ιδεολογικό δόγμα της αμοιβαίας αναγνώρισης όλα τα ε, ένωμα συστήματα των κρατών μελών φαίνεται ότι είναι ίσα. Αυτό όμως δεν είναι ορθό. Είναι θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα εγκρίνει κάποια από τα δοκιμασμένα στοιχεία του αγγλικού νομικού συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεμπρετό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η ποινική δικαιοσύνη ανήκει στην κυριαρχία των κρατών. Γι' αυτό είμαι κατά της πρότασης οδηγίας που θέλει να δημιουργήσει ευρωπαϊκές εγγυήσεις για τα παιδιά τα οποία διώκονται ποινικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι και αλλιώ είναι ανίκανη να προσφέρει τέτοιου είδους εγγυήσεις. Ε, στο άρθρο 6 η πρόταση οδηγίας αναγνωρίζει τα παιδιά στο δικαίωμα του να έχουν δικηγόρο αλλά λέει ότι υπάρχουν εξηγήσει όταν η προστασία από δικηγόρο δεν είναι αναλογικά απαραίτητη και στο άρθρο 12 τους δίνει το δικαίωμα να κρατούνται ξεχωριστά από τους ε, ενηλίκους και ταυτόχρονα προβλέπει την εξαίρεση, λέει ότι όταν δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό ε, έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστρεψε τη Γεωργία, τη Γαλλική, κατέστρεψε ε, τη βιομηχανία τη γαλλική, κατέστρεψε την ε, φύλαξη των συνόρων μας και τέτοιου είδους εγγυήσεις απαράδεκτος που προτείνει θα καταστρέψουν και τη δικαιοσύνη. Η κυρία Μορβάη δεν είναι εδώ, η κυρία Μέτσολα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομη πρόεδρε. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών τα οποία ε, κατηγορούνται έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να την χάνουν τη σωστή προστασίας. Είναι απαραίτητο η εκπαίδευση επίσης των παιδιών ή μάλλον η ενημέρωση των παιδιών να διασφαλιστεί. Είναι απαραίτητο τα παιδιά να γνωρίζουν το τι συμβαίνει και δεν θα πρέπει να είναι απομονωμένα τα παιδιά αυτά μέσα στο νομικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να την χάνουν προστασίας μέσω και της σωστής ενημέρωσης. Και να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μπορούν επίσης να κρατούνται και κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, αλλά θα πρέπει πάντα να μην ξεχνάμε ότι είναι ανήλικοι και γι' αυτό κάθε μορφή προστασίας είναι απαραίτητη. Η οδηγία αυτή αντικατοπτρίζει θα έλεγα τα εθνικά δικαιώματα και θα πρέπει να υποστηριχθεί πλήρως. Μόνικενς. Εξοχότατε επίτροπε συνάδελφοι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα παιδιά ακόμα και κάτω από την ε, ηλικία της ποινική ευθύνη ε, ασκούν παράνομες πράξεις. Ωστόσο πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανήλικοι. Αυτό ισχύει για τις δικονομικές διαδικασίες, όχι μόνο για την απόφαση του δικαστηρίου. Χρειάζεται λοιπόν να τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική συνδρομή από συνήγορο, η ειδική αντιμετώπιση, ατομική αξιολόγηση, η ειδική διαδικασία ερωτήσεων. Επιπλέον τα άτομα, αυτά, τα άτομα που εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές πρέπει να εκπαιδεύονται για να μπορούν να αξιολογήσουν σωστά την κατάσταση σε κάθε φάση της διαδικασίας και τα γενέστερα. Εν τέλει, Υπάρχουν ζητήματα εκπαίδευσης, ε, σχέσεων με οικογένειας, ε, θετική εξωτερική ε, παρέμβαση. Πέραν της ποιότητας μπορεί, δεν μπορεί να υπάρξει ευτυχής παιδική ηλικία. Η δυστυχισμένη παιδική ηλικία είναι αυτή που κυρίως δημιουργεί τους εγκληματίες. Οι κοινωνίες μας πρέπει να βοηθήσει να αντιμετωπίσει αυτές τις πιο ευάλωτες ομάδες εγκληματιών. Η κυρία Ζαμπόρσκα, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μας εκπλήσει και μας απογοητεύει το ότι δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμός για τη δίκαιη δίκη για τα παιδιά. Τα δικαστήρια βασίζονται ε, σε ατελή στοιχεία. 12% των ε, συμμετεχόντων σε ποινικέ διαδικασίες είναι παιδιά. Χρειάζονται ειδικέ διατάξεις για να τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών. Δεν πρέπει τα παιδιά να ε, γίνονται θύματα πολύπλοκων δικονομικών διαδικασιών. Χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής που αποτελεί ένα μέσο ενίσχυσης της δικαιοσύνης, ώστε να μην παρακάμπτεται η δικαιοσύνη. Συγχαίρω επίσης και την εισηγήτρια για την προσπάθειά της να διασφαλίσει τις ειδικέ εγγυήσει για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Nous allons conclure avec... Ευχαριστώ και κλείνουμε με την κυρία Ward. Ένα λεπτό παρακαλώ. Χαιρετίζω την έκθεση που έχει συντάξει η Κατερίνα με την οποία ιδρύσαμε από κοινού ε, την, ε, κοινοβουλευτική, την ομάδα στο Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα των παιδιών. Ε, όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν δικαιώματα σε δίκαιη δίκη όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν δικαίωμα σε δίκαιη αλλά τα παιδιά είναι ιδιαίτερω ευάλωτα. Χαίρομαι λοιπόν που η έκθεση τονίζει ότι θα πρέπει πρώτο μέλημά μα να είναι τα δικαιώματα του παιδιού. Ω μέλο τη επιτροπή για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση τονίζω το ρόλο τη της επανένταξης των παιδιών που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Θα πρέπει να προσφέρονται μέτρα για την εκπαίδευση και για την κοινωνική ένταξη και επανένταξη των παιδιών και των νέων που έχουν ε, περάσει μέσα από το ε, σύστημα ποινική δικαιοσύνης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ε, παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν αποτύχει στο παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης. Ο κύριος Πόσπριλ στο, πλαίσιο του συστήματος Catch the Ο κύριος Πόσπιση, διορθώνω το όνομα, δεν το πρόφερα σωστά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όταν ήμουν υπουργό δικαιοσύνη στη χώρα μου υποστήριξα την ευθυγράμμιση των ε, διαδικασιών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Όπως επίσης στήριξα τα δικαιώματα των νέων παραβατών και κατηγορουμένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να παρακολούθησε τη συζήτηση στην Δημοκρατία της Τσεχίας που προηγήθηκε σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών σε καταστάσεις όπου το παιδί έχει ε, διαπράξει μια σοβαρή πράξη. Δεν θα πρέπει ε, ανήλικοι όταν διαπράττουν κάτι το πολύ σοβαρό όπως φόνο δεν θα πρέπει ε, να υπάρχει ανωνυμία σύμφωνα με την κοινή γνώμη της χώρας μου. ογδόντα έξι παιδιά βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη και όμως μόνο έξι κράτη μέλη έχουν ειδικό εισαγγελέα ανηλίκων. απαιτείται λοιπόν να υπάρξουν ειδικά δικαστήρια ανηλίκων. πρέπει να διαμορφώσουμε την έννοια της δίκαιης δίκης για τα παιδιά. πρέπει να υπάρξει σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού όπως προσδιορίζει και η σύμβαση του οηε. αυτό σημαίνει πέραν των άλλων κατάρτιση των δικαστών αλλά και των ίδιων των δικηγόρων οφείλει λοιπόν κάθε κράτος μέλος να διασφαλίσει συνδρομή δικαστική με δικηγόρο στους ίδιους τους ανηλίκους. ο στόχος πρέπει να είναι η επανένταξη στην κοινωνία πρέπει να είναι η προστασία και όχι η περιθωριοποίηση. δεν θέλουμε ένα σύγχρονο όλιβερ τουίστ και την παρέα του που περιέγραψε ο τσαρλς ντίγκενς στο λονδίνο το. 1838. πρέπει λοιπόν να λάβουμε σοβαρά μέτρα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πρόεδρε. Υποστηρίζουμε αυτό το σχέδιο οδηγία και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εγγυόμαστε αυτά τα δικαιώματα του παιδιού. Δεν θα πρέπει ε, να θίγονται τα παιδιά λόγω της νεαρής τους ηλικίας. Δεν ξέρω αν η ένωμη τάξη στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι οποίοι είναι θύματα μιας εγκληματικής πράξης που διαπράττεται από παιδιά θέλουν ενημέρωση. Δεν είναι τόσο εύκολο λοιπόν το θέμα. Ε, δεν είναι τόσο εύκολες οι λύσεις. Ευχαριστώ κλείνει η διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ και δίνω το λόγο στην Επίτροπο Γιούροβα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Το μόνο που μπορώ να πω κλείνοντα είναι ότι αυτή η οδηγία αποτελεί άλλη μια σημαντική συνεισφορά για τις δικονομικές εγγύησεις για τους υπόπτους ή κατηγορουμένους που έχουν δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Χρειάζονται ελάχιστα πρότυπα και αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμη απουσιάζει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό προτείνουμε αυτούς τους εναρμονισμένους κανόνες. Η πρόταση αυτή δίνει ειδικέ εγγυήσεις για τα πιο ευάλωτα άτομα που είναι τα παιδιά και γνωρίζετε ότι πρόσφατα υιοθετήσαμε την οδηγία για το τεκμήριο αθωότητας και προτάθηκαν και οδηγίες για τις δικονομικές εγγυήσεις και ε, θα προταθεί και η ειδική οδηγία για ε, τη συνδρομή δικηγόρου και για το ευεργέτημα παινίας. Τα μέτρα τα οποία προτείνονται είναι μέτρα τα οποία είναι προς όφελος των παιδιών Μιλάμε για ε, περιπτώσεις όπου το παιδί διαπράττει ε, πράξεις ε, που τιμωρούνται από την κοινωνία. Όμως η κοινωνία δεν θα πρέπει να στερεί το παιδί από την ευκαιρία του να δοκιμάσει μια νέα αρχή στην κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Κινίτσι, θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους και για τις παρεμβάσεις και για την εκτίμηση που εξέφρασαν για την ε, συμφωνία. Ελπίζω να υπάρξει υποστήριξη από τους ίδιους και τις πολιτικές τους ομάδες. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο και για την, ε, την ομιλία της σήμερα και για την τεχνική υποστήριξη. Αύριο θα ψηφίσουμε ένα κείμενο που ε, παρέχει μια σειρά δικαιωμάτων για τους ανηλίκους συμβάλλουμε έτσι στην δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ποινική δικαιοσύνης και το νομικό αυτό κείμενο μαζί με άλλα θα ενταχθεί στην συνολική αρχιτεκτονική των δικονομικών δικαίων, αλλά κυρίως θα έχει στόχο να καλύψει τις διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων από κράτος σε κράτος, λαμβάνοντας υπόψη στην ποινική διαδικασία τα ειδικά χαρακτηριστικά των ανηλίκων, ιδιαίτερα την τροτότητά τους, ιδίως όταν είναι σε δύσκολη κατάσταση, δηλώνοντας ότι τα δικαιώματα των ε, ανηλίκων πρέπει να προστατεύονται ανα πάσα στιγμή. Κλείνω, Πρόεδρε, με μια προσωπική παρατήρηση. Τώρα, φέτος, συμπληρώνονται 20 χρόνια από την εμπλοκή μου στον χώρο της ε, δικαιοσύνη των ανηλίκων. Χαίρομαι λοιπόν που ήμουν εισηγήτρια για ένα κείμενο που θα βελτιώσει τη συνθήκη των, ε, τη συνθήκη των ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ.